εάν το νόμισμα ορισμένων χωρών υποτιμάται θα ακολουθήσουν και άλλα αυτή την πορεία. Ευχαριστώ κύριε Μπρόντς και θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Πρόντι.